Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε όπως πάντα πολύ πυκνό πρόγραμμα. Βέβαια σας καλωσορίζω όλους πρώτα Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Και περνώ αμέσως στην ημερήσια διάταξη και το σημείο 1. Όπως ξέρετε, η ψηφοφορία για τα δικαιώματα των παραγωγών στην ψηφιακή αγορά έχει αναβληθεί για τον Ιούλιο. Στην Ολομέλεια λέω και για τη σημερινή μας ψηφοφορία να δεχθούμε την ίδια αναβολή, αφού η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων έχει κάνει αναβολή μέχρι τον Οκτώβριο, από ό,τι γνωρίζω, άρα έχουμε χρόνο για τη γνωμοδότησή μας. Ε, μπορείτε να δεχθείτε λοιπόν την τροποποίηση αυτή της ημερήσιας διάταξης. Καλώς εγκρίνεται λοιπόν. Και σημείο δεύτερο της ημερήσιας διάταξης, πρακτικά της 25ης Απριλίου. Τα έχετε στα έγγραφά σας. Έχετε αντιρρήσεις για τα πρακτικά όχι. Όπως συνηθίζουμε λοιπόν, εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασής μας εγκρίνονται. Σημείο 3, του Προέδρου και πρώτα έχουμε την διερμηνία σήμερα στις εξή γλώσσες. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, εσθονικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Υπενθυμίζω πάλι, όπως πάντα, ότι γίνεται η μετάδοση μέσω του διαδικτύου της συνεδρίασης και επίσης η αποφάση των συντονιστών της 30 Μαΐου του 2017 απεστάλησαν σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας στις 31 Μαΐου και θεωρούμε ότι εάν μέχρι τις 6 Ιουνίου δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις θα εγκριθούν. Και προχωρώ λοιπόν στις ψηφοφορίες αλλά πρώτα επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για την ε, μεγάλη εκδήλωση για την επέτειο των 30 ετών από το Erasmus Plus στο Στρασβούργο. Είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση πανηγυρική τόσο στην Ολομέλεια όσο και στη συνέχεια στις συζητήσεις που έγιναν σε διάφορα πάνελς και τις διάφορες άλλες εκδηλώσεις που οργανώσαμε στις 13 Ιουνίου ήταν νομίζω ε, μια εκδήλωση ε, με πολύ καλή απήχηση, με πολύ καλή ε, αποδοχή από το κοινό, το οποίο οποία οφείλουμε ιδιαίτερο στο Στέφαν Μάνεφ και το Λούκα Ματιώτη και γενικότερα τη γραμματεία της Επιτροπής μας που έκανε πάρα πολύ σκληρά. Τους ευχαριστούμε λοιπόν όλους θερμά. Πολύ σκληρή δουλειά. Χρειάστηκε πολύ συντονισμός ε, μεταξύ των διαφόρων ε, οργάνων και υπηρεσιών που συμμετέσχουν σε αυτή την εκδήλωση και επιτέλεσαν το έργο τους με μεγάλη επιτυχία οι συνάδελφοι. Η Κορνέλια Κρούζα επίσης, η οποία ήταν αρμόδια για τα θέματα τεών συνεντεύξεων τύπου και ο κύριος Λατίνη από, την, ε, από το επιτελείο του Πρόεδρου Ταγιάννη έκαναν επίσης καταπληκτική δουλειά και συνέβαλαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων, αλλά φυσικά τα συγχαρητήρια πάνε σε όλους τους ε, υπαλλήλου ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε όλο το προσωπικό. Ήταν μεγάλος ο κόπος, το ξέρω, άξιζε όμως τον κόπο. και δίνουμε βέβαια και νέε κατευθύνσει για το Erasmus Plus ταυτόχρονα. Επίση, θέλω να έχετε υπόψη ότι σήμερα το απόγευμα η συνεδρίασή μα θα ξεκινήσει στι 3. Γίνεται μαζί με την ΕΜΠΛ. Στο 4Q1 όμω, 4Q1 σε άλλη αίθουσα, το μέλλον του θεματολογίου για την Ευρώπη και την ε, δικαιοσύνη. Και μετά συνεχίζουμε εδώ με την ακρόαση για τον Brexit. Επίσης, Ευχαριστώ τη Χέλγα Τρούπελ, η οποία αναλαμβάνει για αύριο το πρωί την ε, προεδρία της συνεδρίασης. Και το λέω αυτό γιατί θα γίνει πολύ σύντομη η συνεδρίαση αύριο, άρα αν δεν σας πειράζει. Μια και πρέπει να πάω σε μια εκδήλωση απονομής ε, πτυχίων σε ένα πανεπιστήμιο, είπα να μην το χάσω αυτό όπως είπα είναι μικρή συνεδρίαση. Ε, έχετε όλοι λοιπόν προσκληθεί αύριο πλατεία Λουξ. Το χρυσό περίπτερο. Και ε, εορτασμοί της ημέρας για τους πρόσφυγες με πρωτοβουλία της Helga Trüppel. Προσκαλούνται όλοι οι συνάδελφοι για να ακουστεί δυνατή η φωνή μας και σας παρακαλώ να είστε όλοι αύριο μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας παρόντες σε αυτή την εκδήλωση, στο Χρυσό Περίπτερο, στην πλατεία Λουξεμβούργου. Και τώρα περνώ στις ψηφοφορίες. Τρεις είναι οι ψηφοφορίες που έχουμε για σήμερα. Με πρώτη αυτή που αφορά την ε, ε, πανεπιστημιακή μετεκπαίδευση εξ αποστάσεως ε, σπουδές ως κομμάτι μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διαβίου μάθηση. Ο Σάρθος Βέρ έχει την έκθεση αυτή αναλάβει και τον ε, ερωτώ αν θέλει να πει δύο λόγια πριν την ψηφοφορία. Όχι. Επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ξεκινώντας με την τροπολογία υπαριθμών 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 67. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές. Ας το επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 15 κατά. Απερίφθη. Συμβιβαστική υπαριθμών 9 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 κατά αποχές απερίφθη 78 υπέρ κατά αποχές ας το επαληθέψουμε παρακαλώ 78 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας 14 υπέρ 16 κατά απερίφθη 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 89. Ναι, με περδέψατε λίγο. 89, παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, απεριφθεί. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 97 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά Αποχές απερίφθη. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 ε, συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές ας το επαληθεύσουμε 137 πέρας απερίφθη 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, να επαληθεύσουμε την 138 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 17 ψήφι υπέρ 13 κατά 139 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 140 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 Απερίφθη. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές ας το επαληθεύσουμε 168 πέρας 16 ψήφοι κατά 7 ψήφοι υπέρ 7 αποχές απερίφθη 169 υπέρ Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας το επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 15 ψήφι πέρα, 14 κατά. 170 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ε, επαληθεύουμε την 180. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, 4 κατά. Ε, αν σηκώνατε το χέρι σας θα μπορούσα καλύτερα να καταλάβω που πάει η ψηφοφορία. 181 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ, κατά άποχες. Απερίφθη 189 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 192 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 193 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 195 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 196 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 21 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 207 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές δεν κρίνεται. Συμβαστική 22 ψήφι κατά αποχές δεν εγκρίνεται. Η τροπολογία 214 πέ. κατά αποχές δεν κρίνεται. 215 Υπέ. κατά αποχές εγκρίνεται. 216 Υπέ. κατά αποχές εγκρίνεται. Η σημαστική 23 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 221 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ κατά αποχές Απορρίψετε. 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 228 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. ψηφιπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 15 είπε, Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. Συμβαστική 4 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 19 είπε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 habe oh, Ξέχασα την 20, αν είναι δυνατόν. Για να πάμε λίγο πίσω. 20 λοιπόν. Στη σελίδα την προηγούμενη, είπε. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα θα πάμε στην τροπολογία 28. είπε, Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 30 επέ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 επέ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά τι έγινε. όχι, επειδή εγκρίθηκε η 40 πρέπει να πάμε στη 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 είπε, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 60 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές αυτό μάλλον θέλει έλεγχο γιατί ήταν πολύ μικρή διαφορά αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται 13 υπέρ, 17 κατά. Α, δεν ήταν και τόσο κοντά. 64 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η υπέρ 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απο, ε, εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Okay, okay. Wir haben noch was vergessen. 100. Ah, ξεχάσαμε και άλλη την 101. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Κάπου γλίστρισε και πρέπει να τη βρούμε τώρα. Στη σελίδα 4, μάλιστα. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την τροπολογία 101. Ζητώ συγγνώμη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε λοιπόν το σύνολο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. 24 ψήφοι υπέρ, μία κατά και πέντε αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια θερμά στον εισηγητή και τους σκιώδης. Δείχνει ο που φορείας ότι ήταν πολλή δουλειά, χρειάστηκαν πολλοί συμβιβασμοί, πολλές ε, διαπραγματεύσεις. Συγχαρητήρια λοιπόν. Επόμενο θέμα σχέδιο γνωμοδότησης, κανόνες σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων εφαρμοστεί σε ορισμένε διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Ουφ. Η συγγήτρια είναι η κυρία Πέτρα Κάμερ και μπορούμε να περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία ενδεχομένως να είναι λίγο περίπλοκη. Παρακαλώ την προσοχή σας και τη συγκέντρωσή σας για να μην κάνουμε καμιά στραβή. 123. Έχει αποσυρθεί. Οπότε θα περάσουμε στη συμβαστική 1. Ψήφι Κατά. Α, Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά στο λέξουμε καλύτερα παρακαλώ. Μισοψηφία. Μισοψηφία. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Συμβαστική 2. Ψηφιπέρ. Κατά. Απόχες. Και αυτό θέλει έλεγχο. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 16-14. Προχωρούμε. Η τροπολογία 138 είναι λίγο πιο πίσω, θα τη βρείτε κάποια στιγμή. Υπέρ 138, σελίδα 5 είναι. Στη δική μου, λέει η Είναι αρκετά πιο κάτω. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Συμβαστική 3. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 15-15 ισοψηφία. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό παρακαλώ θα ήθελε έλεγχο. Αρχίζει τώρα. Geschlossen. Πέρας. 19-10 εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Dann gehen wir zu 149. Genau, der fällt nicht. 149 που δεν καταπίπτει. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Τώρα πάμε στο συμβιβασμό 6 υπέρ κατά άποχες και αυτό μάλλον χρειάζεται επαλήθευση αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση και λίγη εγκρίνεται 20-10 178 υπέρ κατά 178. 178 είπα. Περιμένω να τη βρείτε. Μετά το συμβασμό 12, είναι στη σελίδα 14. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας, 13-16 απορρίπτεται. 14, dafür. Συμβαστική 14, υπέρ. Κατά. αποχές. Αυτό θέλει έτσι αλλιώς έλεγχο. Συμβαστική 14 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Να, εγκρίνεται 29-9. Ναι. Τροπολογία 180 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Α, ζητώ συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. Έχουμε και άλλε τροπολογίε. Ε, βιάστηκα. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα η 15 συμβαστική υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 15-15. Οπότε θα πρέπει να τις ψηφίσουμε. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Δεν ψηφίζεται. 184 αρχίζει η ψηφοφορία. Geschlossen. Τέλος. Απορρίπτεται 14-16. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό χρειάζεται έλεγχο. Αρχίζει τώρα. Geschlossen. Mit 16. Απορρίπτεται 12-16. 185 υπέρ κατά αποχές και αυτό παρακαλώ να το ελέγξουμε αρχίζει τώρα η ψηφοφορία Geschlossen. περας το απορρίπτεται 12-18 186 υπέρ κατά αποχές και αυτό παρακαλώ να το ελέγξουμε αρχίζει τώρα η ψηφοφορία και λίγη. Απορρίπτεται 14-16. 187 Είπε. κατά, αποχές. Και αυτό θέλει έλεγχο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και τελειώνει. Απορρίπτεται 12-18. 189. Ψήφι Κατά άποχες. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Αν θέλετε να το τσακάρουμε. 189 παρακαλώ. 189. Πέρασε. Απορρίπτεται. 11, 19. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευσης. Είναι περίπλοκη η ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα λοιπόν η επαλήθευση. Πέρα. Απορρίπτεται. 13-17. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές και εδώ θα χρειάζεται έλεγχος. Για τη συμβαστική 16 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 15-15. Συμβαστική 17 είπε Κατά. Άποχες. Το είχα φανταστεί. Θα χρειαστεί έλεγχος και σε αυτήν. 17 συμβαστική αρχίζει ηλεκτρονική επαλήθευση. 15 15-15 απορρίπτεται. Επίσης. Λοιπόν, θα πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά μία-μία τις τροπολογίες. 193, 194, 195, 196. Είναι όλες Λιπάμε Υπέρ. Κατά. Αποχές. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά χρειάζεται κάθε φορά έλεγχος. Πέρασε εγκρίνεται 16-14. Τροπολογία 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ φωνάζει κάποιος. Ωραία. Να το τσακάρουμε και αυτό. Αρχίζει λοιπόν η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 18 συμβαστική. Πέρας. Εγκρίνεται. 17-13. Τροπολογία 202. Ψήφι Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση. Geschlossen. Mit 12 zu 14 abgelehnt. Απορρίπτεται 12-14. Änderungsantrag 17. Dafür. Η 17 είπε. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. τροπολογία 16. Ψήφι είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19. Είπε. Κατά αποχές, έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για την 19 συμβαστική. Πέρασε. Εγκρίνεται 16-14. Οπότε ακολουθεί η συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές την συμβαστική 20 ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ κατά αποχές έτσι κι αλλιώς θα χρειαστεί έλεγχος πάμε αρχίζει τώρα η ψηφοφορία Πέρασε. Απορρίπτεται 14-15. Συμβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Αν θέλετε μπορούμε και να το ελέγξουμε. Ευχαριστώ. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για τη συμβαστική παρθών 21. Geschlossen. 14 υπέρ 16 κατά απορρίπτεται. Η τροπολογία 26 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 27 είναι στην επόμενη σελίδα. 27 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η ε, 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 32 υπέρ. Που είναι προηγουμένος βέβαια. Συγγνώμη, 37 εννοούσα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη, 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Άποχες αυτό θέλει έλεγχο. Αρχίζει παρακαλώ η ψηφοφορία. Απόρριψε την ισοψηφία 15-15. Ωραία. Προχωράμε. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αρχίζει η ψηφοφορία. 16-17 εγκρίνεται. Η τροπολογία 23. Συμβαστική. Συμβαστική 23. Επέρα. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 14-15. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό χρειάζεται παλήθευση. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά ας το τσεκάρουμε για καλό και για κακό. Αρχίζει η ψηφοφόρη. Τέλος. Απορρίπτεται 14-14. Η τροπολογία 43 επέ κατά αποχές και αυτό χρειάζεται επαλήθευση. Μάλλον έχει εγκριθεί για να δούμε. Αρχίζει ψηφοφορία για τη 43. Να σηκώνετε παρακαλώ τα χέρια σας λίγο πιο ψηλά, αλλιώς δεν ξέρω τι ψηφίζετε. Πού είμαστε τώρα. Συμβαστική 25. Στη μέχρι επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό χρειάζεται έλεγχο. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 15-15. Συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά αποχές και αυτό παρακαλώ πρέπει να επαληθευτεί. Είναι η συμβαστική 26. Πέρασε. 15-15 απορρίπτεται. Η τροπολογία 51. Ψηφί περα Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27. Υπέρ. 27. Συμβιβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα φανταστήκατε ότι πρέπει να το τσεκάρουμε. Αρχίζει η ψηφοφορια Πέρασα. Πέρασε. 15-15 απορρίπτεται. Συμβαστική 28. Μήπως να τα κάνουμε κατευθείαν ηλεκτρονικά, να ξεμπερδεύουμε. Συμβαστική 28, λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρας. 14-16 απορρίπτεται. 60. 60. 60, 61 και 62 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές και αυτό χρειάζεται έλεγχο αρχίζει το ηλεκτρονική ψηφοφορία Geschlossen. Πέρας. 15-15 απορρίπτεται. Dann kommen wir jetzt zu 63 und 64. 63 και 64 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό θέλει έλεγχο. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρας. Απορρίπτεται 14-15. Η τροπολογία 66 υπέρ κατά, αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αν θέλετε να το λέξουμε. 66, αρχίζει ψηφοφορία. Περάς. Απορρίπτεται 14-15. Η 65 έχει αποσυρθεί, συμβαστική 29. Προτείνω να γίνει κατευθείαν ηλεκτρονικά, δεν έχει νόημα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 14-16. Και τη 30 απευθείας ηλεκτρονικά παρακαλώ, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 14-16. Πάμε στι τροπολογίες 69 και 70 τώρα. Ψήφι Κατά. Αποχές. Θέλετε να το ελέγξουμε, παρακαλώ. Νομίζω έχει απορριφθεί. Ισοψηφία 15-15 απορρίπτεται. Η τροπολογία 71 ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά ας το ελέγξουμε και αυτό. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 12-16. Η τροπολογία 72 είπε κατά αποχές απορρίπτεται. Η 73 έχει αποσυρθεί. Η συμβαστική 31 ε, ηλεκτρονικά αρχίζει μέσω η ψηφοφορια Απορρίπτεται 14-15. Συμβαστική 32, επίσης ηλεκτρονικά, αρχίζει ψηφοφορία. Αγκρίνεται 16-13. Τώρα, συμβαστική 33, υπέρ. Κατά. Αποχές και αυτό θέλει έλεγχο. Παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Και λίγη. Εγκρίνεται 15-14. Τροπολογία 83. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Παρ' όλα αυτά να το ελέγξουμε παρακαλώ. Δεν τσεκώνεται χέρια. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Και τελειώνει. Εγκρίθηκε 20 υπέρ, είναι κατάσταση. Το συγγνώμη, αλλά δεν φάνηκε από την ψηφοφορία τόσο σαφώς. Ε, πάμε λοιπόν στη συμβαστική 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος αρχίσει η ψηφοφορια Πέρας. Εγκρίθηκε 16-14. Η τροπολογία 92. Ψήφιπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό θα παρακαλούσα να το ελέγξουμε. Συμβαστική 35 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία και τελειώνει. Εγκρίνεται 16-14. Συμβαστική 36. Ηλεκτρονικά κατευθείαν. Γιατί πάντα τόσο μικρέ διαφορέ. Ε, Μα χίζει η ψηφοφορία. Πέρασε εγκρίνεται 16-14. Συμβαστική 37 και αυτή ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 15-15. Ε, συμβαστική 38 ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 15-15. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το επαληθεύσουμε και αυτό. 100 λοιπόν. Πέρασε. 16 υπέρ, 14 κατά. Ε, 16 κατά, συγγνώμη, 14 υπέρ, απερίφθη, 101 υπέρ, κατά. Αποχές, απερίφθη. Συμβαστική 39, ηλεκτρονικά και πάλι. Αρχίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 40 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απερίφθη. 102, 103, 104, 105 ταυτόσημες μαζί, υπέρ. Κατά αποχές, ναι, πρέπει να το επαληθεύσουμε, λοιπόν Αρχίζει η ψηφοφορία. 102, 103, 104, 105 μαζί είναι. Πέρας. Ε, εγκρίνονται 15 υπέρ 14 κατά. 107 ε, υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά. Αποχές ε, απεριφθεί. 110 υπέρ κατά αποχές 110 λοιπόν επαληθεύουμε ηλεκτρονικά σας παρακαλώ Πέρασε. 14 υπέρ, 15 κατά. Απερίφθη. 108 υπέρ. Κατά αποχές, ας το επαληθεύσουμε και αυτό, 108, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 17 κατά, 9 υπέρ, απερίφθη η 41 και την κάνουμε κατευθείαν ηλεκτρονικά παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 13 υπέρ, 14 κατά, απερίφθη. 42 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται 14 υπέρ, 13 κατά. Συμβαστική 43, ηλεκτρονικά πάλι. Αρχίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 44. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται 15 υπέρ 13 κατά. Συμβαστική 45. Ηλεκτρονικά. Και αρχίζουμε. Πέρασε. Απερίφθη. 46 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απερίφθη. 14 υπέρ, 15 κατά. 120 παρακαλώ, υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη. 121 υπέρ, κατά αποχές απεριφθεί. 122 έχει αποσυρθεί. 15, 15 παρακαλώ υπέρ, κατά αποχές απερίφθη και τελική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 18 υπέρ 9 κατά. Ευχαριστώ. Δύσκολη ψηφοφορία. Και ως εισηγήτρια πρέπει να πω ότι θα πρέπει να επαληθεύσω την κατάσταση και επιφυλάσσομαι να αποσύρω την υπογραφή μου. Θα σας ενημερώσω μόλις μελετήσω το κείμενο. Σιλβία Κώστα. Ήθελα να πω, Πρόεδρε, ότι δεν πρόλαβα να ψηφίσω στην τελική ψηφοφορία γιατί δεν ε, πάτησα το κουμπί πριν την κλείσετε. Ήθελα απλώς να σημειώσω ότι είμαι υπέρ. Ευχαριστώ. Σίλβια, μπορείς σε παρακαλώ να, να επαναλάβεις γιατί δεν σε άκουσα. Κυρία Κώστα. Ναι, απλώς ε, πάτησα με καθυστέρηση το, κουτί, το κουμπί της ψηφοφορίας και δεν κατεγράφει η δική μου ψήφο στο τελικό αποτέλεσμα. Ήθελα να πω ότι υπερψηφίζω. Καλώς λέει η Πρόεδρος και τώρα προχωρώ στην προσεχή ψηφοφορία που αφορά την πρόταση γνωμοδότησης, σχέδιο γνωμοδότησης, έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής κόντ του ελέγχου των προϋπολογισμών σε σχέση με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης ε, κόστους αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Εγγύησης για την Νεολαία με την κυρία Κομοντίνη, η οποία όμως δεν είναι εδώ, αν δεν απατώμε. Ας ψηφίσουμε λοιπόν κατευθείαν και σας υπόσχομαι ότι θα είναι εύκολη αυτή η ψηφοφορία, πολύ πιο εύκολη. Υπάρχει μόνο ένα υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη δύο υπέρ κατά αποχές μάλλον εγκρίθηκε αλλά στο πολυθέψουμε πέρας ζητώ συγγνώμη είχε απορριφθεί δεν μπόρεσα να το δω ε, Υπολογία 3 υπέρ κατά αποχές. Μα να σηκώνετε το χέρι όμως να καταλαβαίνω. Να επαληθεύσουμε λοιπόν. 3. Πέρας. 16 κατά 9 υπέρ απερίφθη, 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 4 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 8 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά. 17, 17. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται απερίφθη. Να επαληθεύσουμε αν θέλετε την 17. Πέρας. Απερίφθη. 18-19 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθεί. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26-27 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 28 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 29 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απερίφθη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 40 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 41 υπέρ κατά άποχες νομίζω ότι εγκρίθηκε αλλά στο επαληθεύσουμε 41 Πέρας. Εγκρίνεται 22 υπέρ, Ζήτω συγγνώμη, αλλά πάλι δεν είχα σαφείς ενδείξει ή εγώ δεν ε, κοίταξα καλά. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 44 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 45 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Και τώρα έχουμε το τελικό, την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, μία ψήφος κατά. Τέσσερις αποχές. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια κυρία Κομοντίνη. δύσκολες οι ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνατε πολύ προσπάθεια. Δεν ήταν εύκολα. Λοιπόν, μπορεί να ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες, αλλά όχι και τη συνεδρίαση. Και γι' αυτό παρακαλώ. Όποιος θέλει να αποχωρήσει από την αίθουσα, να το πράξει κατά το δυνατόν αθορύβος. Σημείο 7 στην ημερήσια διάταξη. ανταλλαγή απόψεων με, τον, με τους εμπειρογνώμονες ε, που προσδιορίζονται στο Συμβούλιο Επιλογής της πόλης που θα γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα. Παρακαλώ ησυχία. Τρεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επιλογή της πολιτιστικής πρωτεύουσας έχουν δώσει την, τον απολογισμό για τις εργασίες 2015-2017. Τους προσκαλούμε λοιπόν στη σημερινή συνεδρίαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω εδώ σήμερα. Σας καλωσορίζω κυρία Σίλβια Άμαν, κυρία Φαρντίνα και κυρία... Να με συγχωρήσετε λίγο στην προφορά. Φλάζε. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ. Επιτροπή Πολιτισμού θα μας ενημερώσετε για τις δραστηριότητές σας στο όργανο αυτό και κυρίως τις μεγάλες προκλήσεις την αξιολόγηση και παρακολούθηση των δράσεων των πολιτιστικών πρωτεύουσών και βέβαια θέλουμε και να μας πείτε πώς βλέπετε το ίδιο το πρόγραμμα. Στη δε προσεχή συνεδρία των συντονιστών θα έχουμε την ευκαιρία ε, να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τους συντονιστές για την παράταση του προγράμματος. Θα δώσουμε λοιπόν στις ειδικού, μόνο γυναίκες έχουμε, να μας κάνουν τι παρουσιάσεις τους και βεβαίως μετά θα μιλήσουν οι συντονιστές και όποιος άλλος συνάδελφος ενδιαφέρεται. Έχετε 4 5 λεπτά στη θέση σας για να μας παρουσιάσετε τις προτάσεις και τις θέσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που έκανατε δεχθεί, δεκτή αυτή την πρόταση και βέβαια για την πρωτοβουλία σας να μας ενημερώσετε εκ του σύνεγγης για τις εργασίες σας Παρακαλώ, ποια από σας θέλει να ξεκινήσει. Καλή σας μέρα. Καταρχήν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Πρόεδρο αλλά και το σύνολο της Επιτροπής Πολιτισμού για την πρόσκληση αυτή και τη δυνατότητα που μας δίνεται να αλλάξουμε απόψεις μαζί σας. Όπως γνωρίζετε είμαστε ε, ε που έχουν ε, οριστεί από αυτή την Επιτροπή ε, το όνομα του Ευρωκοινοβουλίου για να συμμετάσχουμε σε αυτό το πάνελ που θα επιλέξει ε, τις πολιτικές πρωτεύουσες ε, για την περίοδο 2015-2017. Μετά από δύο έτη θητείας μπορούμε πλέον να μοιραστούμε μαζί σας ε, τις ε, εμπειρίες μας. Πιστεύουμε ότι έχει προσθεμένη αξία η όλη διαδικασία, όχι μόνο για την πρόθεση του πολιτισμού στην Ευρώπη, αλλά και για το ευρωπαϊκό ε, σχέδιο γενικότερα. Καταρχήν να συστηθούμε, μια και είμαστε εδώ ως άτομα. Το όνομα μου είναι Κριστίνα Φαρίνια, ε, ζω στο Πόρτο στην Πορτογαλία. Δύο δεκαετίες έχω εργαστεί στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, ε, στην ανάπτυξη πολιτικής, ε, της πολιτικής πολιτικής. Ε, ανάπτυξη επίσης της, συνεργα... συνεργασία πολιτικής και τη διευκόλυνση της κινητικότητας, ε, στη δημιουργία δυνατοτήτων ε, για του επαγγελματίε του κλάδου, την πρόθεση της επιχειρηματικότητα, τη καινοτομία και των νέων αναλλακτικών μοντέλων επιχειρήσεων. Το όνομα μου είναι Σίλβια Αμάν από την Αυστρία, κοντά στο Λίντς, που ήταν η πρώην πολιτιστική πρωτεύουσα εργάζομαι στην πολιτιστική και αστική ανάπτυξη εδώ και πολλά χρόνια. Έχω εμπειρία από ταμία, ταμεία. Ε, επίσης ε, συμμετείχα στο σχέδιο LINS 2009, στο project αυτό, σε ό,τι αφορά το σκέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και επίσης ε, είμαι συμπρόεδρος της ομάδας OMC για την, τον πολιτισμό και της, τη βιομηχανία της δημιουργίας. Δηλαδή ασχολούμαι και με αυτό το ζήτημα. Το όνομα μου είναι Αγνίσκα Βλάζελ. Έρχομαι από την Πολωνία. Έχω οργανώσει πολλές ε, ε πολυτομεακές δραστηριότητες. Ε, επίσης κάνω ένα PhD στην, στο Πανεπιστήμιο του Λίτς ε, στον τομέα των, των, των οπτικοακουστικών Λοιπόν, έχουμε επιλέξει κάποια ζητήματα για τη συζήτηση σήμερα και θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα στις εργασίες του ίδιου του πάνελ και στη συνέχεια θα σας πούμε ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις της νέας απόφασης, ποια είναι τα νέα κριτήρια για τον ορισμό των πόλεων από το 2020 2033, 2023 συγγνώμη, θα δούμε ποιες είναι οι βασικές τάσεις, ε, ποιοι είναι οι παράγοντες επιτυχίας της όλης πρωτοβουλίας και ε, ποιε είναι οι προοπτικέ για το μέλλον. Όπω είπε η Κριστίνα, πρώτα απ' όλα να σα ενημερώσουμε για το έργο μα. Πώ δηλαδή λειτουργεί το πάνελ. Έχουμε φέρει μερικέ εικόνε από την, ε, ε, το πάνελ επιλογή ε, στην Ιρλανδία. Τον Ιούλιο έλαβε αυτή η συνάντηση. Βλέπετε εδώ του εκπροσώπου του πάνελ. Συνήθω είμαστε 10 μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν και εθνικοί εμπειρογνώμονε. Στην προηγούμενη περίπτωση στην Ιρλανδία δεν είχαμε βέβαια, αλλά συνήθω έχουμε έω και δύο εθνικού εμπειρογνώμονε. Υπάρχουν από εκεί πέρα διαχειριστικέ αρχέ, το Υπουργείο Πολιτισμού δηλαδή συνήθω τη εν λόγω χώρα, καθώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι είναι παρατηρητέ, παρακολουθούν δηλαδή ε, και εποπτεύουν έτσι ώστε να ακολουθείτε η κατάλληλη διαδικασία σύμφωνα με την οδηγία και το πλαίσιο που έχει θεσπιστεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιλογή, σε γενικέ γραμμέ μα παίρνει περίπου ένα έτο. Ξεκινάει πέντε χρόνια πριν αναλάβει ε, το, πριν τα απονεμηθεί ο τίτλο τη ε, πολιτικής υπάρχει μια προεπιλογή ε, στην τελική επιλογή ε, και με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε το πάνελ παίρνει την απόφαση και συστήνει ε, μία από αυτές τις πόλεις ε, προς την αρχή διαχείρισης. Όταν λοιπόν επιλέγεται αυτή η πόλη, πλέον το πάνελ παίζει το ρόλο της εποπτείας. Είμαστε κατά, κάποιο τρόπο οι, οι θεματοφύλακες ε, των ε, πολιτικών πρωτεύουσών, δίνουμε συμβουλέ, συνοδεύουμε την όλη προπαρασκευή, διότι έχουμε και πραγματογνωμοσύνη σχετική που θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η στρατηγική, το όραμα τη πόλη αυτή ε, θα διαφυλαχθεί παρά τι αλλαγέ βεβαίω ε, που ε, επιβάλλει πραγματικότητα συχνά στα διάφορα project και βεβαίω η κάθε πόλη έχει τη, τη δική τη διαδικασία Παρακολούθηση και αξιολόγησης. Ε, στην τελευταία συνάντηση, γιατί γίνονται τρει συναντήσεις με τους εκπροσώπους των πόλεων και μια επίσκεψη στην πόλη, στην τελευταία συνάντηση, δηλαδή ένα έτος πριν ε, την, ε, το έτος Πολιτική πρωτεύουσα ε, συζητούμε και ψηφίζουμε και συστήνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όχι να δοθεί το βραβείο Μελίνα Μερκούρη 1,5 εκατομμύρια ευρώ το οποίο δίδεται σε αυτή την πόλη. Ε, στο συνολικό προπολογισμό τη ΕΚΟΚ είναι ένα μικρό ποσοστό. Αυτό ένα μικρό ποσό είναι όμω συμβολικά σημαντικό για την πόλη, διότι αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται, υποστηρίζει, συνεχίζει να υποστηρίζει αυτό το project έω το τέλο και με βάση αυτή την επιβεβαίωση ε, και γίνεται και μια μόχλευση ε, κεφαλαίων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα νέα κριτήρια μετά τη νέα απόφαση για την περίοδο 2020-2033. Ε, το πρώτο είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη της πόλης. Δηλαδή οι πόλεις θα πρέπει να έχουν θεσπίσει, να έχουν εγκρίνει ε, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη της πόλης, όπου βεβαίως ο πολιτισμός ε, είναι πλέον ένα στρατηγικό εργαλείο, παίζει ένα στρατηγικό ρόλο, αλλά όπου και ο ΙΚΟΚ δεν είναι η αρχή και το τέλο ε, πέρα από την πολιτική πρωτεύουσα. Ε, πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια, πρέπει να υπάρξει μια κληρονομιά, αν θέλετε, ε, μετά από το έτος πολιτικής πρωτεύουσα. Το δεύτερο κριτήριο είναι ένα κριτήριο το οποίο είναι οριζόντιο, αφορά το σύνολο του προγράμματο, το σύνολο τη διαδικασία. Είναι η ευρωπαϊκή διάσταση. Όταν εξετάζουμε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, Προφανώς οι πόλεις θέλουν να πάρουν ε, μια θέση στην ευρωπαϊκή ε, αυτή πλατφόρμα. Ε, όταν βλέπουμε τώρα το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε ιδέες, σε έννοιες που να έχουν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, διότι οι πόλεις από εκεί και πέρα ε, θα δουν τι έχουν κάνει άλλες πόλεις για να συνδεθούν και να αναπτύξουν κοινά project ε, με βάση κοινά συμφέροντα και κοινά ζητήματα. Το πρόγραμμα ε, δεν εκπονείται απλά από κοινού, αλλά εκτελείται και παράγεται επίσης από κοινού. Έτσι λοιπόν ε, οι, οι εταίροι είτε είναι άλλες πόλεις ε, που ήταν στο παρελθόν πολιτικές πρωτεύουσες που θα είναι, είτε είναι καλλιτέχνες από άλλες πόλεις, είτε από την Ευρώπη είτε και από αλλού, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο πάντως στο πρόγραμμα και αυτή η κινητικότητα ε, ισχύει ε, αμφίδρομα και προς τα μέσα και, και προς τα έξω. Δηλαδή θέλουμε και να ε, διαφημίσουμε την πόλη στο εξωτερικό αλλά και να προσελκύσουμε ανθρώπους στην πόλη. Ε, δεν βασιζόμαστε μόνο στο παρελθόν βέβαια της πόλης αλλά και στα μελλοντικά project αυτό το πρόγραμμα λοιπόν θα πρέπει να αναφέρεται στην κληρονομιά, στις, παρα, παραδόσεις αλλά και στην καινοτομία, στο νέο όραμα που σχετίζεται, σχετίζεται με τις νέες μορφές ε, τεχνών. Τέλος, ε, το πρόγραμμα έχει ως στόχο και τους επαγγελματίες του κλάδου. Θέλουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε δυνατότητες ε, όχι μόνο για την εφαρμογή του προγράμματος αλλά και για να μείνει κάτι από όλη αυτή τη διαδικασία. Άλλα στοιχεία τώρα τη νέα απόφαση απόφασης 2020-2033 για την περίοδο 2020-2033 είναι το, το στρατηγικό σχεδιασμός ε, για το σύνολο ε, του αστικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, ο πολιτισμός δεν είναι μια απομονωμένη δραστηριότητα που αφορά απλά ένα πολιτιστικό πρόγραμμα ή κάποια καλλιτεχνική δραστηριότητα. Είναι ε, μια ευκαιρία, είναι μια συγκυρία για να υπάρξει μια επένδυση στο σύνολο των υποδομών τη πόλη και αυτές οι υποδομές ε, δεν επικεντρώνονται μόνο στο πολιτιστικό τομέα. Βεβαίω είναι σημαντικό το πολιτιστικό σκέλος πρέπει να συνάδει δηλαδή με το πολιτιστικό και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Παραδείγματο χάρη, να μια πόλη ε, οργανώνει μια μεγάλη έκθεση, θα πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλο χώρο και να είναι διαθέσιμο για την έκθεση αυτή. Ε, υπάρχει και θέμα προσβα... το θέμα τη προσβασιμότητα όμω, ε, την κινητικότητα, όλο και περισσότερε πόλεις ε, επενδύουν στα πλαίσια της πολιτική πρωτεύουσα ε, σε περισσότερα μέσα κινητικότητα ε, πιο φιλικά προς το περιβάλλον ή κάποια σημεία συνάντηση, κάποιες πλατείε πλατείες στις πόλεις. δεν πρέπει να είναι μόνο ένα μέρος διέλευσης, πρέπει να είναι και μέρη, πολιτισμού, που θα λάβουν, να λάβουν χώρα δρόμενα, συζητήσεις, είναι μια πραγματικά ολοκληρωμένη στρατηγική ε, την οποία παρουσιάζουμε όλο και πιο συχνά ε, στις ε, αιτήσει. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, το γνωρίζετε και στα πλαίσια του προγράμματος Creative Europe, η ανάπτυξη του κοινού είναι σημαντικό στοιχείο και αυτό φαίνεται και στα project για την πολιτική πρωτεύουσα. Μιλάμε όλο και περισσότερο για το ποια θα είναι η απήχηση. Ε, πάμε πέρα από ε, την πολιτιστική εκπαίδευση για τα παιδιά ή κάποια συνεργασία με τα σχολεία. Θέλουμε να συμμετάσχουν οι κοινότητες, οι τοπικές, ε, να υπάρχει μια συμβολή στην κοινωνική συνοχή. Ε, ομάδες που δεν είναι ενδεχομένως απολύτως ενταγμένες ε, θα μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερο, καλύτερα. Επίσης, το τρίτο σημείο είναι το θέμα της διαχείρισης μπορεί να μην είναι το πλέον σημαντικό, αλλά είναι εξίσου κρίσιμο. Διότι όταν ένα project δεν έχει τύχη σωστή διαχείριση, δεν βασίζεται σε μια στέρεα χρηματοδότηση, δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να πετύχει. Ε, το είπε και η Κριστίνα, η πόλη δεν βασίζεται μόνο στα 1,5 εκατομμύρια. Υπάρχει, ε, υπάρχουν τα 1,5 εκατομμύρια από το, το βραβείο Μαλίνα Μερκούρη, αλλά ε, μπορούν έτσι να βρεθούν και άλλα κονδύλια από το 2020, ε, από, το, από τα προγράμματα Εράσμους. Ε, οι πόλεις δηλαδή εδώ επενδύουν πολλά, αλλά και οι γύρω περιοχές. Και κάτι ακόμα, εδώ σε αυτή τη διαφάνεια, είναι σημαντικό για να καταλάβετε, θα σας παρουσιάσουμε και μετά, κάθε τρία χρόνια οι υποψήφιες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και πέρυσι επιλέξαμε την πόλη του Νόβισαντ και αυτός ο ανοιχτός χαρακτήρας του διαγωνισμού θα ισχύσει και για το 2024 δεν είναι μόνο τα δηλαδή της Ένωσης λοιπόν ε, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη σε ό,τι αφορά το ECOC ε, της πόλης δηλαδή που, που επισκεφθήκαμε η πρώτη ήταν στην Κροατία στη Ριέκα επελέγει η ΔΙΕΚΑ ήταν 9 υποψήφιες χώρες, ε, τέσσερις ε, πρώτες μέρες προεπιλογής, τελικά κέρδισε η ΡΙΕΚΑ την ψήφο μας. Είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι επικεντρώθηκε στη διευκόλυνση της συμμετοχής ε, η υποψηφιότητα αυτή, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους τοπικούς παράγοντες, αλλά και την, όχι μόνο την, την εθνική, τοπική ηθαγένεια, αλλά και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Προσπαθούμε να συνδέσουμε ε, υπάρχει το σχέδιο 27 γειτονιέ. ε, επίσης ε, υπήρξε μεγάλη ε, εμπιστοσύνη στην ομάδα αυτή ελπίζουμε λοιπόν αυτή η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών να προχωρήσει η δεύτερη πόλη αφορά την Ρουμανία ήταν 14 προεπιλογές, ε, συνέχεια επέλεξαμε 4 ε, και επέλεξαμε την Τιμισοάρα. Ε, μας ε, εντυπωσίασε όχι μόνο ο πολιτιστικό σκέλος, αλλά, αλλά υπήρχε ένα ολόκληρο όραμα το οποίο μοιραζόντουσαν και οι πολιτικές αρχέ εκεί. βασίζεται το όλο project ως μια ιδέα που αναπτύσσεται θα οργανωθεί λοιπόν το πολιτικό πρόγραμμα από κοινού με τοπικές κοινότητες. Δεν είναι απλά δηλαδή παρουσίαση ενός πολιτικού προγράμματος, είναι κάτι το οποίο ε, ξεκινάει από τις τοπικές συζητήσεις. Επιλέξαμε επίσης ε, την Ελλάδα από 14 ε, προεπιλογές και 3 στην τελική φάση. Την Ελευσίνα είναι μια μεσαίου μεγέθους πόλη, όχι μακριά από την Αθήνα, που θα είναι ένα ε, εργαστήριο, αν θέλετε, μιας μεταβιομηχανικής πόλης και πώς αυτή μπορεί να μετατραπεί σε μια πόλη όπου ο πολιτιστικός τομέας θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ε, μετά, στη Λιθουανία, για το 2022, υπήρχαν έξι ψήφιες χώρες, ε, πόλεις, δύο στην τελική περιοχή, τελικά επιλέξαμε το Κάουνας. Εδώ Εδώ έχουμε προγράμματα ε, που έχουν να κάνουν με την, ε, την ε, μνήμη και την σύγχυση, την συνειδητοποίηση, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Να μιλήσουμε τώρα για διάφορες τάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ήδη βέβαια. Οι υποψήφιες πόλεις και οι επιλεγμένες πόλεις είναι όλο και πιο μικρές, η συμμετοχή των πολιτών είναι όλο και πιο έντονη, Επίσης αυξάνεται η συνεργασία ε, μεταξύ των πολιτιστικών πρωτεύουσων. Τα κονδύλια που διατίθενται τη χάνουν σωστής χρήσης και η δημιουργία δυνατοτήτων ε, έχει αρχίσει να γίνεται ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του προγράμματος και έχει απλά ε, μια παρενέργεια. Έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα της συνεργασίας, παραδείγματος χάρη τα τελευταία δέκα χρόνια η οικογένεια των πολιτικών πρωτευουσών συνεδριάζει κάθε χρόνο. Οι νέες πολιτικές πρωτεύουσε ήδη ε, συνεργάζονται, ε, η παραγωγή ε, συνεργάζονται μεταξύ τους σε διεθνές επίπεδο. Πραγματικά θα υπάρχει μια ενισχυμένη συνεργασία όλων των μελλοντικών πολιτικών πρωτεύουσών. Τώρα, κάποιες από τις μελλοντικές πολιτικές πρωτεύουσες ε, βλέπετε εδώ ότι έχουμε χωρίσει τις δύο ομάδες, διότι μετά το 2020 οι πόλεις που έχουν επιλογή, επιλεγεί καλύπτονται από νέα απόφαση. Έχουμε ακόμα την τελική επιλογή του Λουξεμβούργου για το 2022. Κάουνας λοιπόν που έχει ήδη επιλογή και Λουξεμβούργο. Ε, και τώρα προχωράμε προς τα συμπεράσματα. Εμείς έχουμε εντοπίσει κάποιους παράγοντες επιτυχίας, κάποια στοιχεία δηλαδή, τα οποία διαπιστώνουμε όχι μόνο στις πόλεις που κερδίζουν ε, τελικά, αλλά και στις υποψήφιες χώρες ε, ε, και που δεν επιλέγησαν επειδή πρέπει να επιλέξουμε κάποιον. θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για δύο κυρίως στοιχεία. Η καταρχήν η δημιουργία μιας πολιτικής στρατηγικής και η αναγνώριση του πολιτισμού ως ε, στρατηγική πολιτική ε, στα πλαίσια της ευρύτερη ανάπτυξης της πόλης. Για πολλές από τις πόλεις αυτές που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, ήταν η πρώτη φορά που ε, σχεδιάστηκε μια πολιτική πολιτική για την πόλη και αυτές οι πολιτικές εγκρίθηκαν και ισχύουν παρότι αυτές οι πόλεις ενδεχομένως να μην επελέγησαν τελικά. Επίσης ε, υπάρχει αναγνώριση ότι η πολιτική πρωτεύουσα, ο θεσμός αυτός και ο πολιτισμός γενικότερα μπορεί να έχει ε, ε, ευεργετικά αποτελέσματα και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινωνικού, κοινωνικού, κοινωνικής ένταξης. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικού τουρισμού. Θέλουμε να δημιουργούν υποδομές, εκδηλώσεις που είναι ελκυστικές για τους τουρίστες, για τους νέους, για τις επιχειρήσεις, για τους επενδυτές. Ένα κίνητρο και για τους νέους να μείνουν στην πόλη. Επίσης η χρήση του πολιτισμού και των τεχνών μπορεί να βοηθήσει να συνδεθούν διάφορες κοινότητες μεταξύ τους, να, προ... να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη. Δηλαδή ε, είναι ένα μέσο έτσι ώστε ε, διάφοροι άνθρωποι να έρθουν πιο κοντά γύρω από ένα κοινό project. Και ε, φτάνω στο τελευταίο σημείο το θέμα της εταιρική σχέσης και της συμμετοχή. Έχουμε διαπιστώσει ότι σε πολλές από τις υποψήφιες πόλεις για την πρώτη φορά που για πρώτη φορά μάλλον μαζεύουν γύρω τραπέζι διάφοροι φορεί και αυτέ αυτές οι νέες εταιρικέ σχέσεις που δημιουργούνται στη συνέχεια αντέχουν στον χρόνο, μένουν. Ε, αυτό γίνεται σε τοπικό επίπεδο μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών φορέων, πολιτιστικών φορέων, αλλά και με την περιφέρεια και τους ε, γύρω δήμους ε, που συχνά συμμετέχουν ε, στην όλη υποψηφιότητα, αλλά και το εθνικό επίπεδο, διότι είναι ένα εθνικό project τελικά αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Όλοι αυτές τις διασυνδέσεις, όλες αυτές οι ανταλλαγές ε, και αυτά παραμένουν ε, και μετά την, το έτος πολιτικής πρωτεύουσα. Λοιπόν, για να συμβούν όλα αυτά υπάρχουν ε, ακόμα κάποια σκέψεις για το απαιτούμενο πλαίσιο. Εμείς θεωρούμε ότι ένα σημαντικό στοιχείο είναι η χρηματοδότηση από το Creative Europe να συνεχιστεί για την πολιτική πρωτεύουσα κατά την άποψή μας ε, έχει ένα πολύ ε, θετικό αντίκτυπο σε επίπεδο ε, Έχουμε 11 εκατομμύρια από ευρωπαϊκά κονδύλια και μετά έτσι προσελκύονται άλλα 60 εκατομμύρια, προσμένες φορές και περισσότερα. Και βεβαίως υπάρχουν επενδύσεις στις υποδομές και όλες αυτές οι ολοκληρωμένες δραστηριότητε. Θεωρούμε ότι πραγματικά τα χρήματα που επενδύονται πιάνουν τόπο. Υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο. Με το project αυτό η Ευρώπη φτάνει στο τοπικό επίπεδο. Γίνεται αντιληπτή ως κάτι το οποίο οικειοποιούνται οι πολίτες. Τα προγράμματα αυτά ε, σχεδιάζονται κατά τέτοιο, τρόπο ώστε να είναι ολοκληρωμένα, να βλέπουν οι πολίτες, να νιώθουν την Ευρώπη, να έχουν την εμπειρία της Ευρώπης ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, Κατά την άποψή μας, ο θεσμός πολιτικής πρωτεύουσας ε, έχει πολλές και ποικίλε επιπτώσεις σε οριζόντιο επίπεδο, ε, σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό, ε, οδηγεί σε μια καλύτερη ανάπτυξη των πόλεων, οδηγεί σε καλύτερη κοινωνική ένταξη και αυτό θα αντικατοπτρίζεται και στις μελλοντικές στους προγραμματισμούς και στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων ARBECT, ε, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα διαστροτικά ταμεία. Επίσης, τέλος, δεν πρέπει να υποτιμούμε την εικόνα που έχει ήδη σε διεθνές επίπεδο αυτός ο θεσμός της πολιτικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Πρόσφατα ήμασταν σε επαφή με την πρωτοβουλία της πολιτικής πρωτεύουσας Ανατολικής Ασίας ε, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα και Κίνα συμμετέχουν και είναι μια διαδικασία που εμπνεύστηκε από την πολιτική πρωτεύουσα την Ευρωπαϊκή. Ε, είναι λοιπόν ένα πολύ καλό στοιχείο ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ένα περισσότερο, μεγαλύτερο νόημα αλλά και περιεχόμενο σε αυτή την προσπάθεια διεθνοποίησης και για να ενισχύσουμε επίσης τις πολιτιστικές ανταλλαγές και με αυτόν τον τρόπο. Αυτά. Αυτές είναι οι σκέψεις μας για το μέλλον, για τις μελλοντικέ συζητήσεις και αναμένουμε βεβαίως τα ερωτήματά σας. Ευχαριστούμε ήδη εκ μέρους και των τριών που, είχαμε, έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε απόψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα τρία μέλη της Επιτροπής για την ενδιαφέρουσα ματιά που μας άφησαν να ρίξουμε στη δουλειά τους, που μας επέτρεψαν και ε, καταλαβαίνουμε ότι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες έχουν διαχρονική ε, λειτουργία και αυτό που έχει ε, σημασία και για το Κοινοβούλιο δεν είναι να διοργανώσουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια ενός έτους αλλά να αναπτυχθεί ο Δήμος, γενικότερα η τοπική κοινωνία και να συμμετέχει ο κόσμος. Και αυτό το ξεκαθαρίσατε κι εσείς. Ε, και δεν αφορά μόνο τις ε, πόλεις που ε, παίρνουν τον τίτλο της, της πολιτιστικής πρωτεύουσας τελικά, αλλά και για τις υπόλοιπες υποψήφιες πόλεις. Και αυτό το βλέπουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε στις πολιτιστικές πρωτεύουσες. Λειτουργεί στο μεταξύ πολύ καλά αυτό το δίκτυο μελλοντικών και προηγουμένων πολιτιστικών πρωτεύουσων και συνεργάζονται αγαστά με πάρα πολύ ωραία έργα και προγράμματα. Και χαιρόμαστε που επιβεβαιώσατε κάτι που είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και εμείς στις επισκέψεις μας στις πολιτιστικές πρωτεύουσες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή και τώρα θα παρακαλούσα τους συντονιστές να μας πούν αν θέλουν να λάβουν το λόγο. Μισαμπίνε Φερχάιν, θέλεις να πεις τίποτα. Ε, ναι, θέλω. Ε, η Σαμπίνα Φερχάιν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Συγγνώμη που σε διέκοψα κιόλα. Ε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του έργου σας. Μια ερώτηση έχω για τα δίκτυα μεταξύ των προηγουμένων και των ε, επομένων πρωτεύουσων. Είναι λίγες οι πόλεις που συνεργάζονται. Έχετε σκεφτεί να δημιουργηθεί μια συνολική πλατφόρμα για όλες τις πόλεις που έχουν διατελέσει πολιτιστικές πρωτεύουσες και μικρότερες που δεν μπορούν ε, με τις δικές τους δυνάμεις να ε, επιζητήσουν και να αναζητήσουν την ε, συνεργασία για να υπάρξει και μια βιώσιμη συνεργασία και να μείνει και κάτι πίσω. Γιατί Ακριβώς τι είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα, κάτι που διαρκεί ένα χρόνο, τι αφήνει πίσω, τι παραμένει, τι είναι βιώσιμο. Ποιο είναι το δίκτυο, υπάρχει πολιτιστική ανταλλαγή ε, στο Δινεκές, προωθείται γενικότερα στην περιφέρεια, όχι κάτι που συμβαίνει ένα χρόνο και μετά τελείωσε και πάει. και η δική σας Επιτροπή με την επιλογή και την υποστήριξη της συνεργασίας πώς μπορεί ακόμα περισσότερο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε το, πρώτα ένα γύρο ερωτήσεων, θα τις συλλέξουμε και μετά θα απαντήσετε. Η κυρία Τρίπελ, ευχαριστώ και θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση, πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες είναι πραγματικά ένα success story. Έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα στην παιδεία και τον πολιτισμό που ε, ξέρουμε γιατί είναι θέματα με τα οποία ασχολούμαστε ε, ότι φτάνουν στον κόσμο και ανοίγουν τα μυαλά και οι άνθρωποι αισθάνονται περισσότερο Ευρωπαίοι, έρχονται σε επαφή με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι πολλές οι προσκλήσεις και οι ε, προσφορές. πριν από λίγο καιρό πήγαμε στο Όρχους και είδαμε ότι ακριβώς ανοίγει η πόλη, ανοίγουν οι θεσμοί και όχι μόνο, ανοίγουν οι χώροι, ε, έχει ευκαιρία ο κόσμος να ε, περνάει την ώρα του στην πόλη, στο λιμάνι, στο δημόσιο χώρο ε, και ήταν πολύ ωραίο το πνεύμα και η όλη ατμόσφαιρα στο όρους. Yes, I'm, I'm curious what will be... Είμαι περίεργη να δούμε το αποτέλεσμα μετά από κάποια χρόνια ε, υπάρχει μια τάση με κάποιες μικρότερες πόλεις. Είναι θετικό αυτό να βγαίνει στις γειτονιές και σε πιο μικρές πόλεις, σε ε, υπαίθριες περιοχές και να τις διασυνδέεις, αλλά θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Πώς πάει αυτή η προσπάθεια, μπορεί κάποιες πόλεις να έχουν εμφανίσει μεγαλύτερη επιτυχία και κάποιες λιγότερη. Αναφερθήκατε ε, και στις εξωτερικές σχέσεις των πολιτιστικών ε, πρωτευουσών. Τώρα στην Ολομέλη έχουμε την έκθεσή μας για τις ε, εξωτερικές ε, πολιτιστικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θέλετε να το συνδέσετε συγκεκριμένο, διότι ένα θέμα είναι να προωθεί την ιδέα και να τη διαφημίζεις και να λες σε άλλες επίρους τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως θα μπορούσατε πιο συγκεκριμένα να μας εξηγήσετε πώς το βλέπετε αυτό το διεθνές περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητεί κανείς άλλο το λόγο. Γι' αυτό παρακαλώ τις κυρίες του, της Επιτροπής να απαντήσουν όποια θέλει να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας, οι οποίες βέβαια αναφέρονται σε κρίσιμα ζητήματα που μας απασχολούν και μας πολύ συχνά. τα δίκτυα καταρχάς της ΕΚΟΚΣ και πολύ σύντομα. Εμείς θεωρούμε πάντα ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική προσθεμένη αξία και ενθαρρύνουμε όλους τους ε, πολίτες ε, και από αυτό που βλέπουμε, όλες τις πόλεις και αυτό που βλέπουμε από τις πόλεις και τις επαφές που έχουμε περισσότερες όντως μπαίνουν σε αυτού του τύπου τις ανταλλαγές, τουλάχιστον οι πρόσφατα επιλεγήσεις έχουν ε, δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα σε αυτό και βέβαια υπάρχουν και κάποιες νέες ιδέες για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων που μπορούν να αποτελέσουν ένα δρόμο για το μέλλον, αλλά βέβαια θα πρέπει οι πόλεις ίδιες να αποφασίσουν. Εμείς μόνο να ενθαρρύνουμε μπορούμε κατά την ε, διαδικασία επιλογής και κατά την ε, παρακολούθηση να υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία ή να τους προτείνουμε να πάνε σε μια συνεδρία κτλ. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, αλλά το κάνουμε πάντα. Ε, βιωσιμότητα βεβαίως και έχει κρίσιμη σημασία είναι δεν πιστεύω ήδη κάτι το οποίο έχει ενσωματωθεί στην οδηγία που μας διέπει, διότι ε, όλη αυτή η διαδικασία μπαίνει σε μια ε, στρατηγική πολιτισμού, πολιτιστικής ανάπτυξης των πόλεων που κρατάει 10 χρόνια και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προωθηθεί. Βέβαια δεν, μπορούμε, δεν έχουμε αποδείξει αυτή τη στιγμή γιατί το 2020 μόνο ξεκίνησε αυτή η οδηγία να ισχύει, αλλά με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι έχουμε καλύτερη βιωσιμότητα. Και επίσης ε, στοιχεία της βιωσιμότητας απτά που είναι οι υποδομές, ό,τι κατασκευάζεται, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι η παλιάς κοπής βιωσιμότητα. Αυτό που βλέπουμε τώρα σαν νέα εκδοχή, σαν νέα επιλογή των πόλεων είναι πάνω απ' όλα η βούληση να ε, δοθεί δυνατότητα συμμετοχή στον πολίτη, άπαξ και υπάρχει συμμετοχή, άπαξ και υπάρχει αυτή η προσήλωση και η στράτευση σε μια υπόθεση πολιτικής πρωτεύουσα, τόσο περισσότερο διαρκεί ο αντίκτυπο της πολιτιστική πρωτεύουσα και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε και εμείς με τι συστάσεις μας. Για τις μικρότερε πόλεις, Θέλει να συνεχίσει εσύ. Ναι, εδώ έχουμε Πρώτον, το γεγονό ότι ορισμένε πόλει τη Ευρώπη έχουν ήδη αναλάβει πολιτιστικέ πρωτεύουσε στο παρελθόν. Υπάρχουν πόλει που και για δεύτερη και για τρίτη φορά αναλαμβάνουν. Ε, δεν ξανακαταθέτουν λοιπόν μετά. Ε, έχουμε όμω ε, πολιτιστικέ πρωτεύουσε τόσο τη Ρουμανία όσο και τη Ρουμανία που είχαν απλώ τι χειρότερε προτάσει διατυπώσει και έτσι τη Ιρλανδία δεν, μπήκε στην προεπιλογή, της δε Ρουμανίας δεν μπήκε στην ε, τελική επιλογή, γιατί ήταν άλλες προτάσεις καλύτερες. Για τα δίκτυα επίση. Ενθαρρύνουμε όχι μόνο αν ενδιαφέρεται η πόλη να αναπτύξει τις δραστηριότητες με μια άλλη υποψήφια χώρα ή ε, πόλη, ή πόλη που έχει αναλάβει πολιτιστική πρωτεύουσα να γίνει αυτή η διασύνδεση στις επαφές ε, και ιδιαίτερα σε πόλη που έχει αναλάβει πολιτιστική πρωτεύουσα. Ε, αυτέ οι επαφέ έχουν σημασία στι συναντήσει, τα προγράμματα, την ευρωπαϊκή διάσταση που έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολλέ φορέ όσοι είναι το, το μεγαλύτερο ένιγμα για αυτέ. Και επίση τι ε, τις ενθαρρύνουμε να μπουν σε ήδη υφιστάμενα δίκτυα σε θέματα που τις ενδιαφέρουν, είτε πρόκειται για δίκτυα πόλεων, είτε πρόκειται για δίκτυα ε, καλλιτεχνικά, ε, είτε διαφορά άλλα. Συμμετέχουν λοιπόν στα δίκτυα αυτά οι πολιτιστικέ πρωτεύουσε και αυτό μένει ω δεσμό. Και αν μου επιτρέπετε να περάσω εγώ ε, στη διασύνδεση των δύο αυτών θεμάτων, γιατί καθίσταται σαφέ ότι το θέμα δεν είναι μόνο το δίκτυο των πόλεων ως τμήματων της εθνικής διακυβέρνησης και διοίκησης, αλλά των ίδιων των ε, φορέων, των πολιτιστικών και πάνω απ' όλα των ανθρώπων. Και εδώ ακριβώς μπαίνουν οι μικρότερες πόλεις. Και θεωρώ ότι οι μεσές και μικρές πόλεις, προσωπικά θεωρώ, ε, ότι μπορούν να έχουν ακόμη καλύτερο καλύτερη απήχηση στην τοπική τους κοινωνία, πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών τους. Η Τιμισοάρα, παραδείγματι, και η Τρίακα που είχαν αυτή την συμμετοχή, είδαμε πνευματικούς ηγέτες, ε, θρησκευτικούς ηγέτες από κάθε ε, δόγμα και θρησκεία, συμμετοχή των πολιτών σε όλες τις δραστηριότητες, και πάντα βέβαια πρέπει να τονίσετε η ευρωπαϊκή διάσταση, γιατί εδώ ακριβώς ε, έγκυται και η κύρια διάσταση επιλογής για μας. Δεν είναι λιγότερο σημαντικό το θέμα αυτό πλέον. Τώρα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστούν την ευρωπαϊκή διάσταση και να μας πείσουν ότι το πράττουν. Ναι, και αν μου επιτρέπετε κάτι ακόμη για να συμπληρώσω. Βλέπουμε επίσης ότι το γεγονός πως διατυπώνουν τα σχετικά, τις σχετικές προτάσεις οι μικρότερες πόλεις, και έχουν την ε, ικανότητα να αναλάβουν σημαίνει ταυτόχρονα ότι ενώνουν τις προσπάθειές τους ή οφείλεται στο ότι ενώνουν τις προσπάθειές τους για να καταθέσουν την αίτηση. Ακόμη και αν μόνο μία πόλη μπορεί να καταθέσει το σχετικό, τη σχετική πρόταση ε, και αίτηση. Πολλές φορές συνεργάζεται με άλλες πόλεις και διαμορφώνουν από κοινού το πρόγραμμα. Και αυτό είναι μια νέα μορφή κοινου το προγραμμα και αυτο ειναι μια νεα μορφη εταιρικη ε, σχέσεις και συνεργασίας μεταξύ πόλεων. Πολύ σημαντική και πρέπει να την ενθαρρύνουμε. Ναι, να έρθουμε τώρα στις εξωτερικές ε, σχέσεις. Ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητε ε, θα μπορούσαν να αφορούν. Ξέρετε, έχουμε και πολλές ανταλλαγές για γενικότερα ζητήματα στα πλαίσια του πάνελ. Είναι πολύ δυναμική έτσι, η ομάδα μας. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία ε, να πάμε στην Κορέα. Πήγα εγώ στην Κορέα σε μια διεθνή συνάντηση. Είχαμε δύο εργαστήρια που, παρουσιάσαμε στην πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Όχι μόνο η πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης, αλλά την πολιτική πρωτεύουσα όλου του κόσμου. Και συναντήσαμε ανθρώπους από την Ασία που δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή ε, σας είπα προηγουμένως ότι εμπνεύστηκε η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ανατολικής Ασίας από το δικό μας εγχείρημα. Μπορούσαμε να αλλάξουμε απόψεις μαζί τους. Ε, η εμπειρία μας στην Κορέα δείχνει ότι θα μπορούσαμε να επενδύσουμε σε μεγαλύτερη υποστήριξη για την ανταλλαγή πολιτιστικών προγραμμάτων και καλλιτεχνών. Ε, είναι ένας τρόπος αυτός να υποστηρίξουμε και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Πρωτεύουσα, να δημιουργήσουμε διασυνδέσεις, να έρθουμε σε επαφή με αυτές τις άλλες πρωτοβουλίες σε μια πρώτη φάση με την Ανατολική Ασία, διότι εκεί οι χώρες σε κάποιο βαθμό ε, είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία και υπάρχουν στην Κορέα πόλεις παρεμφερα... παρεμφερούς μεγέθους. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ενδεχομένω με κάποια κοινά εργαστήρια αυτό μπορεί να οδηγήσει μεγαλύτερη κινητικότητα μεταξύ των καλλιτεχνών, να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε, εν πάση τη διεθνή διάσταση των προγραμμάτων Ευρωπαϊκή Πολιτική Πρωτεύουσα. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Συζητήσαμε επίση ε, κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα για πιο στρατηγική συνεργασία. Να μάθουμε περισσότερα εμένα από τους δε ε, για το πώς λειτουργούν οι διάφορες πρωτοβουλίες. Από ό,τι φαίνεται αυτές οι ανταλλαγές μεταξύ πόλεων ε, και ένα δίκτυο υποστήριξης πίσω από τις ανταλλαγές ε, θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλος συνάδελφος στο λόγο. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μπάρμπαρα Κέσλερ, τμήματάρχη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν έχει σχόλια ή παρατηρήσει. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πέτρα. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τα σχόλια των βουλευτών και να ευχαριστήσουμε και εμείς τις ειδικού γιατί έχουμε μόνο οι γυναίκες και να τις συγχαρούμε για το έργο τους. Όλα βαίνουν προς την κατεύθυνση που φανταζόμαστε όλοι για το μέλλον των πολιτιστικών πρωτεύουσων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις τρεις σας που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είναι πολύ ωραίο που έχει αλλαγή. Έχουμε τρεις γυναίκες εμπειρογνώμονες που μας παρουσιάζουν το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο σας, για την ενημέρωση ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι προφορίες για το δικό μας έργο. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Στο καλό. So, ich würde jetzt die Sitzung äh, unterbrechen. Διακοπή μέχρι τις 11, όπου ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ. Und den Rest sehe ich äh, hoffentlich um 15 Uhr wieder. Εσάς τους υπόλοιπους ελπίζω να σας ξαναδώ στις 3, στην κοινή συνεδρίαση που έχουμε με την Επιτροπή Απασχόλησης.